Okay, um, welcome. Καλώς σας καλωσορίζω. Ξέρω ότι συμβαίνουν διάφορα δεξιά-αριστερά και είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους να είναι παρόντες ε, στην αρχή της συνεδρίασης. Είχα υποσχεθεί σχετικά με τα benchmarks ότι θα συζητήσουμε το θέμα ή την αναβολή του Είχαμε και άλλα θέματα πιθανότητας αναβολής. Μετά από την ε, αποδοχή λοιπόν της ημερήσιας διάταξης και μία ανακοίνωσης που θα σας κάνω, θα σας προτείνω να κάνουμε μια γενική συζήτηση για τις αναβολές και τι σημαίνουν αυτές. και ποιο είναι το καθεστώς φακέλων τα οποία δεν ολοκληρώνονται, δηλαδή δεν έχει υπάρξει ψηφοφορία επί νομοθετικού ψηφίσματος. Λοιπόν, ας το κάνουμε αυτό. Κύριε Λάγκεν, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. για τη γνωμοδότηση της υποεπιτροπής, της υποεπιτροπής. Κανονικά, αν έχω καταλάβει καλά, την Πέμπτη θα ληφθεί η απόφαση. Αλλά ταυτόχρονα οι πρόεδροι των προέδρων θα είναι σε συνεδρίαση την Πέμπτη, οπότε δεν θα μπορεί να είναι παρόντες. Και μάλιστα η συνεδρίαση δική μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, του Προεδρείου γίνεται στην Πολωνία, οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση παρακαλώ στο Στρασβούργο. Ένα αίτημα ήθελα να σας το καταθέσω. Δεν ξέρω, τώρα βλέπω ότι θέλετε Βέρνερ να συναντιόμαστε Δευτέρα απόγευμα στο Στρασβούργο. Υπάρχει πάντα μία πρώτη φορά. καλός. Νομίζω θα βρεθεί μια λύση κύριε Λάγκεν. Δεν έχω άλλη ανακοίνωση. Λοιπόν, η... για την ημερήσια διάταξη. Κύριος Μίτσελ, έχετε κάνει τεράστια προσπάθεια για το benchmarking και ξέρω πόσο ε, δύσκολο ήταν και σκιώδης. Ξέρω επίσης και τις εκκρεμότητες. Σχετικά τώρα με τα ταμεία των χρηματαγορών υπάρχουν θέματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τεράστιες μετακινήσεις ε, ε, ε, ποσών και αυτό θα ήταν σοβαρό πρόβλημα. Και θα ήθελα λοιπόν σε σχέση με το 5 και με το 7 να αναβληθεί η εξέτασή τους και η αποδοχή, η ψηφοφορία τους. Σε κάποια από αυτά έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, σε κάποια άλλα ε, όχι. Ε, εδώ τώρα κάνουμε μια νομοθετική εμπασπερτώση σοβαρή δουλειά και γι' αυτό ζητώ την αναβολή των δύο ψηφοφοριών του 5 και του 7 έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό όταν πρέπει σοβαρά. Ευχαριστώ Γκέι. Νομίζω ότι οι συζητήσεις που ήθελα να κάνω γύρω από αυτό γυρνούσαν όταν μιλούσα για αναβολεύς. Πράγματι αναφέρομαι στο 5 και στο 7. Κάποια από αυτά τα οποία λέμε ε, ε, είναι μια δυνατότητα. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα κύριε Καντράουι, μην ανησυχείτε. Αφού συζητήσουμε θα αποφασίσουμε. Έχετε το λόγο κύριε Καντράουι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ε, για τα MMF να, γίνουν, να γίνει αναβολή. Υπάρχουν πολιτικές διαφορές, ιδιαίτερα ένα συγκεκριμένο τμήμα της πρότασης. Αλλά έχουμε κάτι μπροστά μας το συγκεκριμένο και θα πρέπει να υπερψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε. Δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι και η διαδικασία, δεν ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία μας, θα πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια, να προετοιμάσουμε εναλλακτικέ προτάσεις, να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει χρόνος για παραπέρα διορθώσεις και γι' αυτό ακριβώς δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει αναβολή για τα MMF. Έχει υπάρξει μια αναβολή Χρειαστήκαμε λίγες μέρες παραπάνω έτσι ώστε να βρούμε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις ευρύτερη βάση. Κατετέθησαν προσυζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα, προδιαθέτουν σε μεγαλύτερη ευελιξία και είναι πιο κοντά στις δικές σας θέσεις, θα έλεγα, παρά τις δικές μας. Και επιμένω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε. Εγώ σας κοιόδη σε αυτή την άποψη έχω. Κοιτάξτε, έχουμε μπει στη συζήτηση για τις αναβολές πριν γίνει η συζήτηση που είχα προβλέψει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνει. Αυτό που ήθελα να πω και θα δώσω στο λόγο στην Έμελη όταν φτάσουμε στα benchmarks. Οι περισσότερες ομάδες έχουν ζητήσει για τα benchmarks αναβολή, για τους δείκτες αναφοράς. Ίσως χρειαστεί να ψηφίσουμε γι' αυτό. Αλλά και σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εκκρεμότητες που έχουμε. Ό,τι δεν έχουμε ολοκληρώσει πριν από το τέλος της πρώτης ανάγνωσης σημαίνει ότι μένει εκκρεμότητα. Και το κοινοβούλιο θα αποφασίσει τι θα κάνει με αυτό. Δεν δεσμεύεται από το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μπορεί φυσικά να δεχθούν την προσπάθεια μέχρι τώρα που έχουμε διανύσει, να ελέγξουν τη συμφωνία υπάρχει επ' αυτής και αυτό θα καθορίσει προφανώς αν θέλουν να αναπέμψουν, αν θέλουν να συνεχίσουν ή οτιδήποτε άλλο. Το νέο κοινοβούλιο έχει κάθε επιλογή δηλαδή ανοιχτή για τη συνέχεια που θα δώσει στα δικά μας μη ολοκληρωμένα. Τώρα, <clears throat> για τους δικούς μου δείκτες αναφοράς, αυτό έτσι κι αλλιώς δεν τελειώνει ποτέ. Εγώ σας υποσχέθηκα ότι θα προσπαθούσα να κάνω κάτι το πάρα πολύ γρήγορο, γιατί και το Συμβούλιο, αν τυχόν το χτυπήσει κεραυνός, θα προχωρήσει και αυτό γρήγορα. Ε, δεν το χτύπησε κεραυνός το Συμβούλιο. Εμείς κάναμε κάποιες προσπάθειες συμβιβαστικές, Φαίνεται ότι ο κεραυνός εμάς φώτισε και εμείς κάναμε κάποια βήματα πρόοδου, αλλά κάποιες πολιτικές ομάδες θεωρούν ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος. Εγώ δεν ξέρω αν θα πρέπει να επανέλθω στις συμβιβαστικές και να τις αναμασάμε συνεχώς. Η δυνατότητα της αναβολής κατετέθη για πρώτη φορά ήδη από τον προηγούμενο Νοέμβριο. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο δύσκολα θέματα εγώ άφησα το βασικό άρθρο χωρίς αλλαγές, αλλά μετά είδα ότι τα θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση είχαν δημιουργήσει περισσότερες δυσκολίες. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της Έμελη, άλλαξα στα πλαίσια της εμβέλειας του τους περιορισμούς τους οποίους είχαμε καταλήξει και στο Στρασβούργο πήγαινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεξιά και αριστερά και εξέφραζε ανοιχτά την ανησυχία της για τον παράνομο τρόπο με τον οποίο εγώ ασχολήθηκα με τα πράγματα έτσι ώστε να σας δώσω στο εσωτερικό ενός κανονισμού τέτοιο περιθώριο ευελιξίας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το κάναμε αυτό και στις κεφαλαιοχές απαιτήσει 750 σημεία έτσι κι αλλιώς επίδειξης ευελιξίας αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι δείκτες αναφοράς είναι πρωτοπόροι, είναι καινοτόμοι, γιατί αλλάζουν κάποιες βασικές αρχές και τους μετατρόπουν σε νομοθετικούς κανόνες και μπορεί κανείς να διερωτηθεί αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μπει καλύτερα στις, σε μια οδηγία και μπορούμε να ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία να μας πει αν κάτι τέτοιο γίνεται. Αν ξεκινήσω από άσπρο χαρτί πάλι, από λευκό χαρτί πάλι, θα πρέπει να σας ζητήσω να προχωρήσουμε γρήγορα σε ένα κανονισμό με κρίσιμους δείκτες αναφοράς. Αυτό θα μπορούσαμε να το προλαβαίναμε στην παρούσα εντολή και να σπρώχναμε και το Συμβούλιο και ίσως να καταλήγαμε σε μια οδηγία η οποία ίσως να μας απαιτούσε περισσότερο χρόνο αλλά θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες διαφορές και τον μεγάλο αριθμό των δικτών αναφοράς. και σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχουν οι αρμόδιες αρχές και η ΕΣΜΑ ε, και κατά πόσον κάποιοι τέτοιοι δείκτες μπορεί να μην χρησιμοποιούνται κτλ. <clears throat> Αυτό είναι ένα θέμα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό ακριβώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο αίτημα για την αναβολή ε, ζήτησε μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, ασφάλεια. Λοιπόν γενικά έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε γρήγορα στους δείκτες αναφοράς. Ίσως να ξαναδοκιμάσουμε. Αλλά πάντως δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ψηφίσουμε πράγματα τα οποία δεν θα υποστηριχθούν και από μεγάλη πλειοψηφία στο εσωτερικό μας, γιατί αυτό είναι ένα μη μήνυμα στους διαδόχους μας καλύτερα να πούμε στους διαδόχους ότι εμείς δεν τα καταφέραμε, προσπαθήστε εσείς. Αν όμως καταλήξουμε σε κάτι το οποίο στηρίζεται από μεγάλη πλειοψηφία, τότε αξίζει τον κόπο και πρέπει να ψηφίσουμε. Γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το επόμενο κοινοβούλιο. Αν όμως το υπερψηφίσουμε με πάρα πολύ ε, πολυδιασπασμένο και λίγο αναρχικό τρόπο τότε σε αυτή την περίπτωση και δεν θα εξυπηρετήσουμε το μήνυμα το τελευταίο που θα δώσουμε και σύν της άλλης δεν θα είναι καθόλου υποβοηθητικό για το επόμενο κοινοβούλιο. Λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα για τους δείκτες αναφοράς. Να μην τους ψηφίσουμε σήμερα, και να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε μια πλειοψηφία που να υποστηρίξει τις αρχικές προτάσεις. Δεν αξίζει τον κόπο να ψηφίσουμε νομίζω σήμερα. Ε, ίσως κάποια θα έπρεπε από τα σημεία αυτού του θέματος των δικτών αναφοράς δηλαδή να συμπεριληφθούν σε μια οδηγία θα πρέπει να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε όταν στα πλαίσια της επόμενης κοινοβουλευτικής εντολής το θέμα τεθεί σε τριμερή διάλογο να ρυθμιστεί και το θέμα αν θα είναι κανονισμός, οδηγία ή κάτι άλλο. Λοιπόν, κάποια από τα σχόλιά μου έγιναν κατανοητά και αφορούν κυρίως το τι ε, οδηγίες θα δόχουμε εν πάση περιπτώσει στους διαδόχους μας. Και σε σχέση με το 7 έχουμε επίσης διαιρέσεις, θα δούμε. Αν ψηφίσουμε όταν ψηφίσουμε. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε πάντως είναι να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μια συνενετική λύση και αυτό θα το πετύχουμε εφόσον έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Η Έμιλη. Εφόσον δεν ψηφίζουμε σημαίνει ότι ε, έχουμε κάποιο χρόνο. Η Έμιλη, ευχαριστώ. Μια που είπε ήδη ότι συμφωνείς για την αναβολή, θέλω να συνεχίσω από αυτό το σημείο κι εγώ. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε, από την πλευρά μας τουλάχιστον, να κλείσουμε τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Εγώ συμβουλεύτηκα και τη γραμματεία επ' αυτού, γιατί ο σκοπός δεν είναι να βγει από την ημερήσια διάταξη. Θέλουμε να δούμε μήπως 3 Μαρτίου μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Επίσης, όταν ζητάς αναβολή, αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνεις τη δέσμευση να κινηθείς πολύ γρήγορα στη συνέχεια ότι θα επανέλθουμε δηλαδή και εμείς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο προκειμένου να έχουμε νέες προτάσεις. Πήραμε τα παραρτήματα την προηγούμενη εβδομάδα. Τα κοίταξαν 22 σελίδες, κανονισμός. Συντάσσουμε κανονισμό και σημαντικό μάλιστα. Είχα την αίσθηση λοιπόν ότι υπήρχαν κάποια κενά, υπήρχαν κάποια σημεία που δεν ήταν τόσο συνεκτικά μεταξύ τους, οπότε μπορείς να μας πεις... Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να πούμε πιο συγκεκριμένα ποιο είναι το εύρος, το πεδίο εφαρμογής. Το θέμα της ΕΣΜΑ μας απασχολεί. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Είναι δύσκολο ο συμβασμός, αλλά πρέπει να τον πετύχουμε ή με τι άλλο να ψηφίσουμε από πλευράς αρχής. Εμείς που είμαστε νομοθέτες θα το καθορίσουμε. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα σημεία κλειδί. Δεν θέλω να μπω περισσότερο σε λεπτομέρειες. Αυτοί πάντως είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους θέλαμε και εμείς την αναβολή. Επίσης βρεθήκαμε με την ομάδα εργασίας και θέλαμε να συζητήσουμε τι θα ψηφίσουμε την Παρασκευή Μόνο όμως πήραμε τον κατάλογο ψηφοφορίας, οπότε μας ήταν πολύ δύσκολο, ήταν δύσκολο να τους εξηγήσουμε τι θα ψηφίζαμε ακριβώς. Οπότε καλό είναι να γίνει αυτή η αναβολή και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα σε επόμενες δύο εβδομάδες. Και να το κλείσουμε όμως το θέμα σε αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ναι και εγώ το ελπίζω. Γιατί όπως έχω πει και κατά το παρελθόν προσπάθησα να συμπεριλάβω τις τροπολογίες όλων και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή τα παρερτήματα είναι συσσόρευση παραρτημάτων και τροπολογιών που έχετε προτείνει. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα καινούριο. Και πάλι προσπάθησα να συμπεριλάβω όλες τις προτάσεις σας. Να έχουμε όμως υπόψη μας ότι από τη μια μεριά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να βγουν ένα σωρό πράγματα από το πεδίο εφαρμογής, ε, αγαθά, ενέργεια και ένα σωρό άλλα πράγματα και από την άλλη έχουμε αυτούς που δεν θέλουν να βγει τίποτα. Είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να συνεπάρξουν αυτές οι δύο θέσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σοφά. Ε, μιλήσατε, λέει ο κύριο Λάμπετ, όταν είπατε ότι είναι καλό να έχουμε ευρεία πλειοψηφία και να περάσει με ευρεία πλειοψηφία η νομοθεσία αυτή. Σωστά αντιλαμβάνομαι ότι για τους δείκτες αναφοράς μπορούμε να πετύχουμε ισχυρή πλειοψηφία. Μπορεί κάποιοι να μην είναι ικανοποιημένοι, αλλά υποθέτω θα είναι 2 τρίτα 1 τρίτο ή 3 τέταρτα 1 τέταρτο, που εγώ θεωρώ ότι είναι ισχυρή πλειοψηφία. Θα μπορέσει δηλαδή να περάσει και να χρησιμοποιηθεί και στην επόμενη θητεία ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα, κατά τα άλλα, οι πρόσφατες εξελίξεις με απασχολούν γιατί βλέπετε Άλλο είναι να θέλουμε να πετύχουμε μια ευρεία πλειοψηφία καλή την πίστη, αλλά όταν ακούω κάποιους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων να λένε πρώτον ότι δεν θέλουν 3% κεφάλαιο πάφερ προστασία ή λίγο πολύ δηλαδή λένε ότι δεν θέλουν τελικά νομοθεσία, ότι θέλουν status quo. Εγώ αυτό δεν το λέω διαπραγμάτευση καλή την πίστη. Και δεν είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε με την πρότασή της. Δεν είναι τυχαίο που πολύ σημαντικοί παράγοντες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Τζίκος κλπ. είπαν ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα κεφάλαια της χρηματαγοράς με μια περίοδο παρατήρησης τριών ετών και μετά να αποφασίσουμε αν θέλουμε phase out ή buffer. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Συνεπώς, εγώ ευχαρίστω, είμαι διατεθειμένος να διαπραγματευτώ καλή την πίστη, αλλά αν κάποιοι άλλοι θέλουν να κάνουν καθυστέρηση και μόνο, τότε πρέπει να το κλείσουμε εδώ και να σταματήσουμε. Παρακαλώ. Η κυρία Μακάρθη. Ναι, και εμένα μου φαίνεται λογική η προσέγγιση που προτείνεται για τους δείκτες αναφοράς. Μερικές φορές όταν προσπαθούμε να πετύχουμε συμβασμούς, και να καλύψουμε τις επιθυμίες όλων, τελικά καταλήγουμε σε μια κατάσταση που ένας είναι ευέλικτος και όλοι δεν είναι. Στις εσωτερικές συζητήσεις που είχαμε στην ομάδα μου φάνηκε ότι μπορεί να λειτουργήσει αλλά δεν είναι σαφές. Πρέπει να υπάρχει νομική σαφήνεια για το τι ζητάμε και όταν εγώ το διάβασα κατάλαβα ότι θα μπορούσε να ερμηνευτεί και αλλιώς. Ότι δηλαδή μπορεί κανείς να ζητήσει από την ΕΣΜΑ εξαιρέσεις. Δηλαδή δεν ξέρουμε τελικά ακριβώς ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής. Είναι δύσκολο να ξεκαθαριστούν αυτά τα ζητήματα λοιπόν και δεν είναι εύκολο να αποφασίσουμε. Πρέπει όμως να αποφασίσουμε αν θέλουμε οδική κανονισμό γιατί δεν μπορούμε να τα μπερδέψουμε και τα δύο. Δεν μπορούμε να ε, συντάξουμε ένα κανονισμό που να μοιάζει με οδηγία. Ούτε μπορούμε να πούμε σε αυτόν ο οποίος καλείται να εφαρμόσει τους κανόνες να διαλέξει. προσπαθούμε να πετύχουμε συμβιβασμούς και στην προσπάθεια αυτή αφήνουμε να περάσουν και κάποιες ασάφειες και δεν πρέπει. Γιατί είναι μια σημαντική υπόθεση και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε για τους δείκτες αυτούς μια πολύ μεγάλη ακρόαση και αν δείτε σήμερα τους Financial Times αναφέρονται στη χειραγώγηση της αγοράς και αυτά τα οποία λένε είναι τελικά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που είχαμε συζητήσει εμεί στην ε, ακρόασή μας για 3,5 δισεκατομμύρια την ημέρα όσον αφορά το Λίμπορ. Συνεπώς δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτούς μας να διατηρηθούν οι ασάφειες αυτές. Όπως ε, είπατε, δεν πρέπει να υπάρχουν ε, μεγάλες διαφορές, κάποιες ομάδες να είναι κατά και στην Ολομέλεια να έχουμε μεγάλες τροπολογίες που θα υποβληθούν. Όχι, η υπόθεση αυτή αξίζει τον κόπο μια καλύτερη μεταστέ. Στο τέλος της θητείας μας πρέπει να έχουμε μια καλή επίδοση. Όπως λέει και η ομάδα μου και αντιπρόεδρος της ομάδας μου, θα βρούμε ένα επικοδομητικό τρόπο να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό στην τρέχουσα θητεία. Ευχαριστώ. Ο Ζαν Πολ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επανέλθω στην αναβολή γιατί αποφασίστηκε και ευχαριστώ. Κατά τα άλλα, δεν πρόκειται απλώς για μια αναβολή έτσι επειδή βολεύει. Πρέπει να ξαναδουλέψουμε το κείμενο. Υπάρχει το νομικό θέμα του κατά πόσο θα πρόκειται για κανονισμό η οδηγία πρώτα απ' όλα. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε κανονισμό. Γιατί τώρα τελευταία με κανονισμούς δουλεύουμε στα οικονομικά. Οπότε αν θέλουμε να εναρμόνιση πρέπει να την πετύχουμε μέσω ενός κανονισμού και όχι να εισαγάγουμε και πάλι ασάφειες. Όσον αφορά τώρα τα αριθμισμένα αγαθά, το είπε και η Αρλίν, το υπενθύμησε, θα έχουμε θα έχουμε το Forex που είναι και κάτι πιο βαρύ από το Libor. Εγώ συνήθως είμαι υπέρ της ΕΣΜΑ, παρόλο που στην αρχή είχα πολλές επικρίσεις, δεν νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε στην ΕΣΜΑ που δεν τη ζητάει ευθύνες που έχουν να κάνουν με το πρώτο επίπεδο. Από αυτή την άποψη λοιπόν διαπιστώνω ότι σήμερα όλοι θέλουν να δώσουν πολλές εξουσίες στην ΕΣΠΑ χωρίς όμως να δώσουν ούτε το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται ούτε τους πόρους, τους οικονομικούς που χρειάζεται. Τι να την κάνουμε μια αρχή για την οποία μετά θα λέμε ότι δεν έκανε τη δουλειά της γιατί δεν της δώσαμε τα μέσα να κάνει τη δουλειά της. Όχι γιατί δεν μπορούσε αλλά δεν της δώσαμε εμείς τα μέσα να το κάνει. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Όπω λέει και η Ερλίν Μακάρθη, καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να κάνουμε καλή δουλειά, παρά για να πούμε ότι το ψεφίσαμε χωρί να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. 3 Μαρτίου, εντάξει, μπορεί να είναι μια ενδεικτική ημερομηνία, αλλά να μην είναι κάτι το απόλυτο. Θα δούμε ανάλογα με το πώ θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ελπίζω το δικό μου κείμενο να ήταν καλύτερο. Ο Δάνα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση έχω να κάνω για να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Γκοζές. Στην αρχή μιλήσαμε για το Λίμπορ και τα άλλα σκάνδαλα. Τώρα βλέπουμε σκάνδαλα στο χρηματιστήριο. Και ένα χρηματιστήριο θα έπρεπε να είναι φοβερά διαφανές. Δηλαδή οι συναλλαγές σε ένα χρηματιστήριο να είναι απόλυτα διαφανείς. Είναι το ελάχιστο. Και εδώ μιλάμε για ένα μικρό τμήμα υπόψη. Διότι έχουμε ένα διάφανο σύστημα και πρέπει να παραμείνει διάφανο. Πρόεδρος. Ωραία. Ελίζα. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι. Πιστεύω και εγώ ότι είναι σημαντικό να αναβληθεί η ψηφοφορία για τους δείκτες αναφοράς και να έχουμε ε, μεγάλη και ισχυρή πλειοψηφία. Τώρα για τις ημερομηνίε. Αν είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό στο νομικό μας έργο να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Δεύτερον, δεν κατάλαβα τελικά αναβάλουμε και τις χρηματαγορές ή όχι. Εγώ δεν βλέπω γιατί. Δεν βλέπω δηλαδή να ισχύουν τα ίδια επιχειρήματα και στο θέμα των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς όπως και στους δείκτες αναφοράς. Οπότε, τι προτείνετε. Πάντω, στην νομοθετικό έργο συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να πάμε όσο γίνεται πιο μακριά για να καθορίσουμε όσο γίνεται καλύτερα τη θέση μας. Πρόεδρος, αυτό που είπα είναι ότι θα αναβάλω τους δείκτες αναφοράς. Ζητήθηκε για τις χρηματαγορές, η συγκητής είναι από τους σοσιαλιστές και έχει διαφορετική άποψη. Σιλβί. Ναι, ούτε και εγώ θέλω να παρατείνω περισσότερο τη συζήτηση. Η δουλειά που έκανε ο συγκητής μας, η συγγήτρια μάλλον, είναι πάρα πολύ μεγάλη βέβαια και είναι σημαντικό να έχουμε ευρεία συνένεση. Υπάρχει πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει. Πρέπει να στοχεύσουμε σε μια ευρύτερη πλειοψηφία. Βρισκόμαστε πάνω σε ένα θέμα στο οποίο δεν υπήρξε απλά ένα λάθος. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά παρανόμησαν. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Θα συμφωνήσω με τον Ζων Μακάρι να το έκανε η ΕΣΜΑ αυτό, αλλά αυτό σημαίνει ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει δυνατότητες τις οποίες δυστυχώς δεν έχει. Λοιπόν, έχουμε πάντως τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε στη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Καλώς, αυτά έχουμε για τα benchmarks. Ο κύριος Μίτσελ, κοιτάξτε, για τους δείκτες αναφοράς πράγματι δεν πρέπει να βιαστούμε αν δει κανείς το πώς νομοθετούμε στην παρούσα φάση, τότε πραγματικά οι ευρωσκεπτικιστές δεν θα ήταν ε, περιθωριακοί αλλά κυρίαρχοι. Εγώ αν έχω τέτοιου είδους ας πούμε κεφάλαια στη χρηματαγορά και βλέπω τον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει κανείς έτσι και σε σχέση με τα σύναψη. Νομίζω ότι ε, φοβάμαι ότι πάρα πολύ λίγοι θα μπορούσαν να στηρίξουν το παρόν σύστημα. Από την άλλη προτείνουμε να το αλλάξουμε, αλλά να το αλλάξουμε με έναν τρόπο χωρίς να γνωρίζουμε σε βάθος περί τίνος πρόκειται. Πράγματι λέμε ότι γύρω στα 400 ε, δις στα MFF, τα οποία θα μπορούσαν πράγματι να προσπαθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε θετικά. Από ό,τι φαίνεται ο κίνδυνος είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αλλάζουμε εμείς την νομοθετική ρύθμιση που ισχύει για όλα αυτά τα κεφάλαια της αγοράς χωρίς να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Αν υπάρχουν προβλήματα συστημικού κινδύνου αν τότε ας έχουμε κάποια τέλη ρευστότητα, ας έχουμε ε, κάποιους άλλους ε, τρόπους ελέγχου και για τα σύναψη και για όλο του είδους τέτοια κεφάλαια. Το θέμα είναι ότι όταν εμείς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και παίρνουμε αποφάσεις, ο κόσμος μας κοιτάει και αναρωτιέται γιατί βιάζονται. Ρόλος μας είναι να έχουμε τον χρόνο που απαιτείται να μην είμαστε πρόχειροι σε αυτά που κάνουμε. Και για τους δείκτες αναφοράς και για τα αμοιβαία κεφάλαια και για τα δύο παρακαλώ αναβολή. Ευχαριστώ. Okay. Να πω κάτι για τα κεφάλαια της χρηματαγοράς. Είναι ένα θέμα για το οποίο πολλές φορές την αλήθεια δεν τη γνωρίζουμε. Και σε σχέση με τις διαβουλεύσεις για τα FSP που γίνονται στην παρούσα φάση, όπου ακούγονται για κάποιες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες περιμένουν την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο βέβαια, από ό,τι φαίνεται σε σχέση με τις κεντρικές τράπεζες, δεν είναι απόλυτα κοινωνές μεταξύ τους σε σχέση με το τι γίνεται στο IFMD και στο usage. Υπήρξαν εκπλήξεις ε, όταν ε, είχαν ενημερωθεί οι μεν για το τι επιθυμούν οι δε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα συμβεί όταν ε, η κατάσταση αυτή, η συζήτηση αυτή καταλήξει σε τριμερή διάλογο. Ελπίζω να υπάρξει περαιτέρω έρευνα από πλευράς των κεντρικών τραπεζών ποια είναι η θέση τους για όλα αυτά τα θέματα. Πάντως η κατάσταση είναι ρευστή, αλλάζει συνεχώς, υπάρχουν ανησυχίες και το βασικό ένστικτο ε, των κεντρικών τραπεζών είναι να μην φύγουν τα λεφτά. Ε, αυτή είναι το βασικό αν θέλετε ε, ρεφλέξ που έχουν οι κεντρικές τράπεζες. Το θέμα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τα σύννεφ τουλάχιστον είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η παρούσα κατάσταση και στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο για όλα αυτά τα ταμεία και για τις καταθέσεις θα πρέπει να γίνει μια κάποια συζήτηση διαφορετική. Αν εμείς πιέσουμε κάποια από τα χρήματα αυτά των ταμείων να θεωρηθούν ως καταθέσεις, τότε δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Φιλίπ έχει ζητήσει εκ νέου το λόγο. Γκέι, σέβομαι αυτά τα οποία ε, λες γενικά, αλλά νομίζω ότι ξεπέρασες τα όρια. Αυτό το οποίο λες τώρα είναι να πετάς αριθμούς δεξιά-αριστερά για να φοβίζεις τον κόσμο. Και αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Στην ουσία ε, ε, κάνεις προσπάθειες εκφοβισμού γιατί λες μην κάνουμε αυτό γιατί θα βλάψει την οικονομία και μην κάνετε το άλλο γιατί δεν ξέρετε τι θα πάει η οικονομία και σύν της οι νομοθέτες που είμαστε εμείς είμαστε ανίδεοι για να μην το πω χειρότερα λέει ο μιλητής. Ε δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν αυτό δεν είναι παρά πολύ μακριά από την αλήθεια. Αν υπάρχει έτσι υπάρξει απόφαση από την SRB ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στο καθεστώς ε, των Ισίνοψ, αυτό είναι κάτι ε, το οποίο το προτείνουμε γιατί ξέρουμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα ή αυτοί οι οποίοι εν πάση περιπτώσει διορίζονται από τους νομοθέτες και από τους άμεσα δημοκρατικά εκλεγμένους ε, γνωρίζουν λιγότερα από αυτούς τους οποίους διορίζει η βιομηχανία του χρήματος. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν τρομοκρατούμε από τον κλάδο αυτό το χρηματοπιστωτικό. Και το να λες ότι όσοι δεν ακολουθούν τις απόψεις της βιομηχανίας είναι ανίκανοι και άσχετοι, αυτό είναι πραγματικά υβριστικό. και δικαίωμα απάντηση, Κοιτάξτε, δεν θέλω να μου δώσει κανένα συμβουλές. Παρακαλώ ψυχραιμία. Εγώ δεν θέλω να είναι τόσο πρόσωπο παγής η συζήτηση. Φιλίπ και εσύ ήσουν <coughs> πολύ στοχευμένος. Ο Γκέι στα σχόλια που έκανε ήταν αρκετά προσεκτικός. Ξέρω Φιλίπ ότι το δικό σου στυλ είναι διαφορετικό. Και πολλές φορές το χρησιμοποιούμε το στυλ σου προς όφελος της Επιτροπής. Αλλά λίγος περιορισμός παρακαλώ στα εκφραστικά σας μέσα. Πράγματι έχουν ακούσει διαφορετικές προτάσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι μόνο η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα που προτείνει. Έχεις δικαίωμα απάντησης, Γκέι. Κοιτάξτε, δεν θα αντιδράσω. <clears throat> Εγώ θυμίζω τη δουλειά μου σαν ομοθέτης ε, ε, είναι κάτι το οποίο εγώ θα κρίνω πώς θα το κάνω. Δεν θα μου το υπαγορεύσει κανείς, ούτε η βιομηχανία, ούτε κανείς άλλος μας ζητήθηκε να ψηφίσουμε κάτι εδώ για το οποίο δεν ξέρουμε. Είναι η αλήθεια τώρα για το, το ότι δεν γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις. Μόνο χρόνο ζητώ να δοθεί ώστε να μπορέσουμε να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η βιομηχανία. Και εδώ και τα, τα ευρωπαϊκά οικονομικά αφορώνται, τοπικές αρχές, πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί επενδυτές ε, αφορώνται άμεσα. Και εδώ πρόκειται για το πώς θα λειτουργήσουν αυτά σωστά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, γιατί στο συμπέρασμα να μην ψηφίσουμε σήμερα καθόλου. Εγώ ζητώ να κάνουμε το έργο μας ως νομοθέτες, να έχουμε χρόνο να το κάνουμε αυτό και να εξετάσουμε τις επιπτώσεις αυτών που συνεπάγονται όλα αυτά τα οποία εξετάζουμε. Είναι το μόνο σημείο που ήθελα εγώ να αναφέρω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Think. Πρόεδρος, όλοι όσοι ήθελαν να παρέμβουν μπόρεσαν να το κάνουν ξεκινήσαμε για, με το θέμα της ψηφοφορίας. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αναβληθεί το θέμα αυτό. Και τα benchmarks, ε, οι βέλτιστες προδιαγραφές ε, θα αναβληθούν. Τώρα να δούμε αν θα αναβάλουμε και τα θέματα τα οικονομικά όσον αφορά τα κονδύλια που εμπλέκονται. Αν αυτή είναι η επιθυμία σας, μπορούμε να ψηφίσουμε διανατάσεως των χειρών να δούμε ποιοι είναι εκείνοι που επιθυμούν να αναβληθεί αυτό το θέμα σε ιστερότερη συνεδρίαση προς ψήφιση. Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά με τις κάρτες μας, για να είμαστε σίγουροι. Εντάξει. Who are you vote? After Louisa. Oh, right, well, we cancel out then. Okay. okay. you. Do Who, who's without a card? Me. Jean Paul. Jean Paul has a point of order. Διαδικαστικό εσύ Jean Paul. Je voulais qu'il soit clair. Ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Εξέφρασα τη θέση μου για αυτό που συζητάμε, αλλά το βασικό ζήτημα στην υπόθεση αυτή είναι <clears throat> ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ΣΥΝΑΒ και τα ΒΙΝΑΒ. Αυτό είναι το βασικό οι σταθερές, δηλαδή καθαρές αξίες ενεργητικού και οι κυβερνόμενες ε, καθαρές αξίες ενεργητικού. Πριν να αρχίσει η συζήτηση είπαμε ότι το θέμα έπρεπε να το ξαναδούμε. Είναι τόσο περίπλοκο που ανάλογα με το πώς θα ψηφίσει η Επιτροπή μας για το ένα ή για το άλλο σημείο, μετά θα υπάρξουν διάφορες επιπτώσεις στο κείμενο. Έτσι όπως έχει σήμερα το πράγμα, και εδώ βέβαια δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν γιατί ο εισηγητής δούλεψε σκληρά και τον ευχαριστώ, αλλά δεδομένου ότι το ζήτημα είναι τόσο δύσκολο, οι θέσεις τις οποίες μπορεί να καταλήξουμε ψηφίζοντας σήμερα θα είναι χωρίς συνοχή μεταξύ τους μερικές φορές. Οι θέσεις μας δεν θα αλλάξουν για το κατά πόσο θέλουμε να διατηρήσουμε τα συνάβη όχι και κατά από ποιες συνθήκες, αλλά αν μη τι άλλο να φροντίσουμε να έχουμε ένα κείμενο πιο συνεκτικό, μια που είναι δύσκολο το θέμα, πάνω στο οποίο δούλεψαν τόσο γραμματεία όσο και συγκητής. Πρόεδρος, η πρόταση δηλαδή είναι να αναβληθεί, όπως είπαμε βέβαια και για τους δείκτες αναφοράς, όχι ΙΣΑΗ, να το αναβάλουμε μέχρι να είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Ωραία, μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Πρώτα απ' όλα για τους δείκτες αναφοράς, γιατί ε, θα το ζητήσουν οι σοσιαλιστές, έτσι δεν είναι. Πρόεδρος, όχι, συγγνώμη. Εννοούσα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, γιατί για τους δείκτες αναφοράς συμφωνήσαμε αμόφανο ότι θα αναβληθεί η ψηφοφορία. Τώρα ψηφίζουμε για το κατά πόσο είμαστε υπέρ της αναβολής. Ναι, σημαίνει ότι είσαστε υπέρ της αναβολής, έτσι. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άλλος ένας δεν έχει ψηφίσει. Α, πέρας της ψηφοφορίας. Αναβάλλεται λοιπόν, γιατί είχαμε 23 ψήφους υπέρ και 15 κατά. Οπότε. άλλο ένα. Παρακαλώ, ο κύριος Ελκαντραουή. Πρόεδρε, φυσικά και σέβομαι την απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής μας. Όμως, Βάσει του πνεύματος των όσων είπε ο κύριος Γκοζές, είμαι έτοιμος να αναβάλω την ψηφοφορία για λίγο. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε να ψηφίσουμε, τόσο το καλύτερο. Και στο μεταξύ μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Στο τέλος όμως πρέπει να υιοθετήσουμε την άποψή μας, τη θέση μας για τα σύννεψη και φαντάζομαι ότι αυτή δεν θα αλλάξει μέσα στις επόμενες μέρες. Οπότε ας συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι είναι η τελευταία αναβολή και ότι την επόμενη φορά θα ψηφίσουμε πράγματι. Έχουν όλοι τις τροπολογίες, έχουν όλοι τον κατάλογο ψηφοφορίας. Μένει να αποφασίσουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ναι. Βερκάρτ. Πρόεδρε, σήμερίζομαι και εγώ απόλυτα αυτά τα οποία ο εισηγητής ανέφερε. Ότι δηλαδή τώρα θα πρέπει το δυνατόν ταχύτερα να ψηφίσουμε, να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Χρειάζεται κάποιο χρόνο για να δούμε ήρεμα, νυφάλια, τον πίνακα κατάλογο ψηφοφορία. Θέλω να επισημάνω, έχουμε μια συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα σε σχέση με το ΕΛΚ, όπου πολλά μέλη από τη δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή συμμετέχουν και θα έλεγα δεν θα ήταν ευνοϊκό αν αυτή την εβδομάδα, την πέμπτη γινόταν αυτό. Σίγουρα είναι ανοιχτό για, όλα τα άλλα, για όλες τις άλλες υποθέσεις, αλλά αυτή την πέμπτη θα ήταν δύσκολο για αυτή την υπόθεση για μας. Πράγματι, συμφωνήσαμε ότι δεν θα είχαμε αυτή την πέμπτη οτιδήποτε. Και δεν έχω και καμιά πρόθεση με τόσο σύντομη, σε τόσο σύντομη προθεσμία να έχουμε θέματα ψήφισης όταν υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Θα επανέλθουμε στο θέμα και θα το ξαναδούμε όταν θα υπάρχει χρόνος διαθέσιμος από την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Αυτό θα σημαίνει ότι ίσως θα πρέπει να δούμε κάποτε τη Δευτέρα να βρούμε χρόνο στο Στρασβούργο στην περίοδο συνόδου. Λυπούμε γι' αυτό, Βέρνερ. Εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Δεν θα έχουμε λοιπόν ψηφοφορίες. Όσοι προσήλθατε για να ψηφίσατε μπορείτε πάλι να αποχωρήσετε. Δεν θα έχουμε ψηφοφορίες. Γι' αυτό τώρα μπορούμε να επανέλθουμε στα κανονικά σημεία της ημερησίας διάταξης 3 και 4. Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για μητρικές και θηγατρικές εταιρείε σε διαφορετικά κράτη-μέλη, διαφορετικών κρατών μελών. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν παρακαλώ να αποχωρήσουν ήρεμα, χωρίς φασαρία. Και θα μπορέσω να δώσω και τον λόγο στη συνέχεια στον συνάδελφο κύριο Νίτρας. Α, εντάξει, όχι, όχι, ο κύριος ε, Κεκούς θα είναι που θα λάβει τον λόγο. Κούκατς. Αν αποχωρείτε παρακαλώ να το κάνετε γρήγορα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Πολύ σας ευχαριστώ λοιπόν. Όταν θα είσαστε έτοιμοι λοιπόν Σας ευχαριστώ κύριε Σάρον Μπόουλς. Ησυχία παρακαλώ. Έχουμε παρεμβάσεις. Δεν πρέπει να φωνάζουν όσοι έχουν τον λόγο. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη από πλευράς Μότσα γιατί δεν παρίσταται σήμερα και έχει και πολύ σοβαρούς λόγους διότι έφερε στον κόσμο παιδί και δεν μπορεί να παραστεί η κυρία Μόιτσα. Θα ήθελα να παρουσιάσω τώρα τα θέματα τα οποία ε, αφορούν ε, την υπόθεση του σχεδίου έκθεσης. Το Κοινοβούλιο είχε λάβει θέση σε σχέση με το θέμα της ε, καταπολέμησης των διαφορετικών εδρών και ουσιαστικά ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα των υβριδικών ε, καταστάσεων όσον αφορά τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα μεταξύ των κρατών μελών καθώς και επίσης να καταθέσει να υποβάλει μια πρόταση για την αναθεώρηση την ε, μεταρρύθμιση του κοινού φορολογικού καθεστώτος ώστε να μην υπάρχει διπλή φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αλλαγές που εισάγονται από την ε, Επιτροπή βρίσκονται στο τραπέζι τώρα και είναι πραγματικά καλοδεχούμενες αυτές οι αλλαγές. Για τα υβριδικά αναντίστοιχα θέματα υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής ε, ο εισηγητής. Και έχουμε κράτη-μέλη τα οποία εφαρμόζουν διαφορετικά καθεστώτα όσον αφορά υβριδικά δάνεια σαν αποτέλεσμα αυτά αντιμετωπίζονται ως ε, ε, δαπάνες που μπορούν να εκπέσουν του φόρου και έχουμε και τα θέματα της ε, κατανομής ε, των ε, κονδυλίων από την άλλη πλευρά. Η ανάγκη αυτή του να αποφύγουμε διπλή φορολόγηση πρέπει άμεσα να καλυφθεί. Η πρόταση που έχουμε στο τραπέζι τώρα η, λαμβάνει υπόψη και τις, τα θέματα που είχαν αναφερθεί το 2010 και σε σχέση και με την φορολόγηση στην πηγή. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως αυτή η εναλλακτική λύση πρέπει να υπάρξει δυνατότητα προσαρμογών. Επίσης, ο κανόνας, η ρήτρα αντιμετώπισης καταχρηστικών καταστάσεων σε σχέση για παράδειγμα με εταιρείες όταν προσπαθούν μέσω μεσολαβητών να επενδύουν κάποιες εταιρείες στα κράτη-μέλη και να δούμε το τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα η εισαγωγή ενός ε, δεσμευτικού υποχρεωτικού κανόνα σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει τα κράτη-μέλη μέσω τέτοιων τεχνητών ε, συμφωνιών ε, να ρυθμίσουν τις δυνατότητες έκπτωσης από την φορολογία πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα και η τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου προτείνεται η ενδυνάμωση του ορισμού μιας μητρικής εταιρείας και το τι θα πρέπει να γίνεται για την αντιμετώπιση του, της τρέβλωσης του, του ανταγωνισμού. Επίσης εισάγεται ένα, ε, το καθεστώς ε, που θα πρέπει από πλευράς ε, φορολογίας των κρατών μελών να μην είναι χαμηλότερο από 75% στα κρατημέλη. Και η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ήδη το 2011 υπεστήριξε αντίστοιχες προτάσεις όταν είχαμε θέματα που παρουσιάστηκαν με αντίστοιχη έκθεση στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Και θα πρέπει όχι μόνο να υποστηριχθεί αυτή η πρόταση αλλά και να υποστηριχθεί και από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πορεία αυτή. Προσβλέπει λοιπόν η εισηγήτρια σε περαιτέρω συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές και τους άλλους συναδέλφους στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστούμε. Δεν γνωρίζω τώρα από πλευρά του ΕΛΚ ποιος θα λάβει τον λόγο. Δεν παρίσταται ο συνάδελφος Ε, τότε λοιπόν η Σιλβή παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Σάρων. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που για καλούς λόγους βέβαια λείπει. Ευχαριστώ και τον αντικαταστάτη της. Θα πρέπει να δούμε κάποια τεχνικά θέματα, αλλά αυτά είναι τεχνικά όπως είπα, λεπτομέρειες. Όχι. Ανησυχώ όταν βλέπω ότι διαβουλεύεται κανείς με το κοινοβούλιο μας για τέτοια θέματα δημοσιονομικά και γίνονται κάποιες συζητήσεις αλλά είναι περιορισμένες οι δυνατότητές μας. Οι συνθήκες αυτό μας επιτρέπουν να κάνουμε. Θα πρέπει να δούμε ακριβώ ποιο είναι το επίπεδο συμμετοχή στο κεφάλαιο. Η συγητή περνάει από το 10% στο 15%. Το ποιο είναι το σωστό ποσοστό δεν ξέρω να σα πω. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και σε σχέση με το νόμιμο επίπεδο επιβολής σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσον όρο. Εγώ δεν είμαι κατά του να υπάρξει ένας κάποιος ανταγωνισμός και ο ανταγωνισμός αυτός να ελεγχθεί κάπως. Το θέμα είναι ποια είναι η πραγματικότητα του επίπεδου επιβολής. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει ε, υπάρχουν κάποιες φορολογικές διευκολύνσεις και δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για νόμιμο μέσο όρο επιβολής, μέσο επίπεδο επιβολής ή για κάτι το διαφορετικό, για πραγματικό, για ουσιαστικό επίπεδο, ε, ε, ποσοστό επιβολής. Λοιπόν, <clears throat> ε, θα πρέπει να δούμε τώρα στα τεχνικά, όπως είπα, θέματα, κάποιες λεπτομέρειες, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει θέμα. Περνάμε λοιπόν τώρα στο Φιλίπ Λαμπέρτς. Με το στυλ που με χαρακτηρίζει όπως είπατε, Πρόεδρε. Έχετε έναν πάρα πολύ έτσι κομψό τρόπο να βρίζετε τον κόσμο, Πρόεδρε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είστε. Καταρχάς να εκφράσω τις ευχές μου στην ε, εισηγήτρια Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν σε σχέση με την λεγόμενη επιθετική φορολογία. Είχα πάει στην Γενική Διεύθυνση ΚΟΜΠ γύρω από τέτοια θέματα. Είναι αλήθεια βέβαια ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν και πάρα πολύ ενθουσιασμό σε σχέση να ακολουθήσουν τους μέσους όρους όπως λέγεται στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα από τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον επιθετικό φορολογικό προγραμματισμό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αν ενθυμούμε από την έκθεση Giggold, είχαμε πει ότι δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το 75% του ε, επίπεδου του επισήμου το οποίο επιβάλλεται. Και αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουμε πάντα και υποστηρίζουμε και τις τροπολογίες του εισηγητή γενικότερα, της εισηγήτριας. Ε, ελπίζω να βρεθεί μια κάποια πλειοψηφία γύρω από αυτό στο Κοινοβούλιο. Ανεξάρτητα από τις απόψεις που έχει ο καθένας για το επίπεδο της φορολογίας, Νομίζω να υπάρξει μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ μας ότι το φορολογικό σύστημα θέλουμε να είναι <coughs> δίκαιο. Να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν την ελευθερία να παίζουν το ένα φορολογικό σύστημα εναντίον του άλλου να ευνοούνται σε σχέση με τις μικρομεσαίες. Εμείς δοξάζουμε τις ε, μικρομεσές γιατί είναι αυτές που γεννούν θέσεις απασχόλησης κτλ. Κι όμως ε, αυτές οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, ε, επιφορτίζονται το βάρος της εταιρικής φορολογίας, φορολόγησης. Και <clears throat> θα πρέπει να πάρουμε ό,τι μέτρο χρειάζεται έτσι ώστε και οι μεγάλες επιχειρήσεις να πληρώσουν το δικό τους ποσοστό και να μην τηρούν μόνο το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου. Θα σταματήσω εδώ. Θα στηρίξουμε λοιπόν την προσπάθεια της εισηγήτριας, θα συζητήσουμε το θέμα με όλους τους εμπλεκομένους και ελπίζω να καταλήξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργη. Ευχαριστώ Σάρων. Μάλιστα. Από ότι εμείς βλέπουμε η κατεύθυνση είναι σωστή σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως με την προσθήκη από πλευράς του συναδέλφου για την ελάχιστη φορολόγηση τουλάχιστον κατά 75% ε, του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας ε, για τις εταιρείες αυτές ε, από τα κράτη-μέλη. Είναι σωστή η πρόταση και την υποστηρίζουμε ρητά. Αποκινούμε την πρόταση που προτείνεται για το άρθρο 1α για την αποφυγή της ε, μη φορολόγησης το θεωρούμε θετικό. Ωστόσο θέλω να επισημάνω σε αυτό το σημείο στο γερμανικό φορολογικό δίκαιο υπάρχει μια, ένα αντίστοιχο αίτημα όμως γενικά έχει διατυπωθεί ώστε να είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό θα περιμέναμε από τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τα στοιχεία σε σχέση με τις ε, επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος να βρίσκονται σε συγκρίσιμο επίπεδο με τα στοιχεία της επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να αποφύγουμε την μη ε, φορολόγηση. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα όσα εκπονήθηκαν από την Κάτω Βουλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλύτερο από ό,τι ισχύει ε, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, δεν επαρκεί η πρόταση αυτή, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ευρέως αυτά τα φαινόμενα. Μόνο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Όταν τα κράτη-μέλη οδηγούνται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση φορολόγησης των επιχειρήσεων που δρούν στην επικράτειά τους. Έτσι τα κέρδη μιας επιχείρησης θα μπορούν μέσα σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ως βάση να φορολογούνται. Και θα μπορούσε να μετρηθεί το κέρδος ε, με τις ε, ε, επιχειρηματικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη και θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε την μη φορολόγηση. Μια τέτοια έννοια φορολόγηση ναι μες ναι, στο πρόγραμμα δράσης του ΟΣΑ αναφέρεται σε σχέση με το shifting όμως θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να υλοποιηθούν. Σίγουρα ένα τέτοιο σύστημα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει βράχη πρόθεσμα με αυτόν τον τρόπο. Όμως από την άλλη πλευρά η ε, σωστή, η δίκαια φορολόγηση για τις ε, πολυεθνικές εταιρείε ε, είναι πολύ δυσχερής υπόθεση. Φτάνουμε στα όρια των δυνατοτήτων μας και από την άλλη πλευρά έχουμε και εξειδικευμένους νομικούς που συμβουλεύουν αυτές τις επιχειρήσεις πόρο απέχουμε λοιπόν από το να επιτευχθεί ένα τέτοιο σύστημα. Από την άλλη πλευρά όμως φαίνεται αυτή η οδηγία να είναι ένα σωστό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση και γι' αυτό υποστηρίζουμε αυτό το εγχείρημα και με τις τροπολογίες που καταθέτουμε. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδηση συγκήτρια μας δεν είναι εδώ. Έχω όμως να ρωτήσω κάτι. Διότι κοίταξα τις τροπολογίες και θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δυνατόν να υπολογιστούν αυτά τα 75% φορολόγησης επί των επιχειρήσεων. Γιατί η φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι τόσο περίπλοκη στις χώρες μέλη. Εγώ ασχολήθηκα για καιρό με αυτό το θέμα και έμαθα ότι σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά είναι υψηλότερα, αλλά υπάρχουν τόσες παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις κτλ. που τελικά η πραγματική φορολόγηση είναι πιο χαμηλή από άλλη χώρα όπου το ποσοστό φορολόγησης αρχικά είναι πιο χαμηλό. Οπότε ρωτάω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδομένου ότι είναι τόσο περίπλοκος ο υπολογισμός. Μπορεί να τον κάνει. Κατά τη γνώμη μου θα είναι αδύνατο να εφαρμοστεί αυτό που προτείνεται εδώ. Προηγουμένως όμως θέλω να ρωτήσω την Κομισιό να μου πει είναι σε θέση στις 28 χώρες μέλη να μας πει ποιος είναι τελικά ο πραγματικός συντελεστής φορολογίας των εταιριών με όλες αυτές τις εξαιρέσεις που ισχύουν. Πρόεδρος, άλλος κανείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ, οπότε θα, θα αναφερθείτε στους φορολογούμενους. Για απαντήστε, αν μπορείτε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή για την επικοδομητική έκθεση που υπέβαλε και τις καλύτερες ευχές μας και συγχαρητήρια για την κυρία Συγήτρια, για τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία ανεφίσαν εδώ και για το, ε, κανονικό, τον μέσο όρο φορολόγησης ε, των ε, επιχειρήσεων που σύμφωνα με τα όσα είχαν προταθεί θα είναι 17,3-17,4% Υπάρχουν κράτη-μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν μειώσει αυτό τον συντελεστή αναέτος κατά μία ποσοστία μονάδα. Όταν κάνουμε λόγο για 17,4% αυτό θα σήμαινε ότι έξι κράτη-μέλη θα πρέπει να αυξήσουν το ποσοστό φορολόγησης ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να ευθυγραμμιστούν όπως ζητεί και η τροπολογία του Κοινοβουλίου. Και είναι γεγονός ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει η φορολόγηση εισοδήματος με ενιαίο τρόπο ε, σε σχέση με αναλογικότητα ε, σε σχέση με τα κράτη-μέλη και να δούμε σε σχέση με τις ε, θηγατρικές εταιρείες το τι μπορεί να γίνει. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι και κέρδη στην ίδια χώρα θα πρέπει να φορολογούνται με το ίδιο ποσοστό 17,4% για έξι κράτη-μέλη θα πρέπει να εισάγεται ένα ε, αντίστοιχο ποσοστό φορολόγησης ε, ώστε να ευθυγραμμίζονται με αυτή την αρχή. Παρότι καλωσορίζουμε ε, την αρχή αυτή, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να δει κανείς πώς μπορεί να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να προβούν σε τόσο ευρύ, ευρύες μεταρρυθμίσεις των εθνικών του συστημάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, θέλετε να επανέλθετε εξ ονόματος ε, της εισηγήτριας. Ευχαριστώ Σάρων. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ε, για τις παρεμβάσεις στη συζήτηση. Και θα έχουμε και την δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια πρόταση. Υπάρχει όμως ευρεία πλειοψηφία υποστήριξη και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Άστριντ, δεν δόθηκε απάντηση στο ερώτημά μου. Δεν μιλάω για το νομιστικό επίπεδο. Για το πραγματικό μιλάω. Μετά από όλες τις δυνατότητες μειώσεων, εκπτώσεων κτλ. Γι' αυτό ρώτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να το καθορίσει. Λόγω των τεράστιων διαφορών στα εθνικά φορολογικά συστήματα, είναι αδύνατο για κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα και για κάθε είδους διαφορετικό τομέα, από τις μικρομεσαίες μέχρι τις πολυεθνικές, να υπολογίζει κανείς ένα ουσιαστικό ποσοστό φορολογίας επιβολής ή θα πάρει κανείς ένα πρότυπο ε, επιχείρησης και θα ε, συγκρίνει κανείς ε, το αποτέλεσμα της εφαρμογής των εθνικών ρυθμίσεων ή θα ακολουθήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει η ενοποιημένα φορολογική βάση εφόσον υπάρχει αυτή η κοινότητα και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα το να επιβάλλει κανείς μετά ένα επίπεδο φορολογίας το οποίο να έχει κάποιο νόημα. Τώρα υπάρχουν διάφορα φορολογικά μέσα εκπτώσεις, δυνατότητες αποκλήσεων, εξαιρέσεων, έμεσων πληρωμών, μπόνους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να τα λάβει κανείς υπόψη του στον καθορισμό. Καλώς. Λοιπόν, ε, θα επανέλθει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι τα πράγματα όμως στο Συμβούλιο πηγαίνουν με αργή ταχύτητα και η απάντηση και στην ερώτηση της κυρίας Λούλεγγ είναι ότι είναι πολύ δύσκολο εφόσον υπάρξει τουλάχιστον ένα, μια κοινή φορολογική βάση τότε τα πράγματα πάνε κάπως πιο γρήγορα. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 25 Φεβρουαρίου, 5 <clears throat> το απόγευμα. Θα τα συζητήσουμε τα θέμα αυτό πάλι στις 17 Μαρτίου και θα ψηφίσουμε στις 18 Μαρτίου. Ελπίζουμε να φτάσουμε στη δεύτερη ολομέλεια του Απριλίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Γιατί είναι αλήθεια ότι η συγγήτρια έχει πάρα πολλή δουλειά, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου οι τροπολογίες παρακαλώ. Περνάμε τώρα στο 4 την ένταξη, την συμμετοχή, την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 23ης Ιουλίου για την κατάργηση της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αναφέρεται στην επανεξέταση της συμφωνίας σε σχέση με την διπλή φορολόγηση. Πρόκειται λοιπόν για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης όταν έχουμε ε, κέρδη τα οποία σημειώνονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Πρόκειται για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για την συμφωνία αυτή αυτό είναι το αντικείμενο. Ε, βλέπουμε ότι τα θέματα αυτά επανεξετάζονται εκάστοτε και σε σχέση με την ένταξη νέων κρατών μελών. Πρόκειται και για ε, το τι μπορεί να γίνει επιδιαιτητικά ώστε η δυνατότητα διπλής φορολόγησης να αποφεύγεται μέσα στο πλαίσιο για παράδειγμα κερδών που σημειώνονται μεταξύ ε, συνεργαζομένων επιχειρήσεων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Η λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής ε, αγοράς ε, διευκολύνεται και διευκολύνονται οι δραστηριότητες διασυνοριακά των επιχειρήσεων και η ένταξη της Κροατίας σε αυτή τη συμφωνία είναι φυσικά σαν απόρρια της ένταξης της Κροατίας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, της πράξης ε, προσχώρησης. Ε, με την προσυπογραφή της πράξης προσχώρησης η δυνατότητα διατησίας είναι υποχρεωτική διαδικασία και η απόφαση αυτή ε, μεταβιβάζεται στο Συμβούλιο μετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτή τη φάση διαβούλευσης ακριβώς βρισκόμαστε και σε αυτή την ε, νομική πράξη που δεν την χάνει οποιασδήποτε αντίρρηση ή αντίδραση ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από την Κροατία. Μια τροπολογία όμως ε, θέλουμε να κατατεθεί και πρόκειται για μια διευκρίνηση απλά και μόνο για την τροποποίηση των διατάξεων της συμφωνίας που τότε θα αρχίσουν να ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή που θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα από το Συμβούλιο ε, η πράξη αυτή. Έχει άλλες προτάσεις στο Συμβούλιο που αναδρομικά ε, μπορούν να έχουν ίσως σαν αποτέλεσμα και μια παράταση του, της διαδικασίας. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο στην Κροατία να προσαρμόσει τις νομικές της πράξεις ε, διαδικασία διαιτησίας. Εμείς πιστεύουμε ότι κατά την τελευταία σύνοδο του Απριλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση αυτή πρέπει να εγκριθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Είναι πράγματι ένα πολύ τεχνικό θέμα. Ο εισηγητής Πάντως εξέτασε καλά την υπόθεση και ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, αρχή της θέσης και νομίζω ότι οι προοπτικές είναι πολύ καλές, με ικανοποιεί και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πρόεδρος Ραμόν. Ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Λέει ο κύριος Τρεμός Εμπαλσέλτς. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Συμφωνούμε με την τροπολογία του εισηγητή του κύριου Νίτρες όλες οι χώρες έκαναν το ίδιο κατά το παρελθόν. Τώρα λοιπόν που έχουμε και νέα χώρα μέλος και συγχαρητήρια για την προσχώρηση αυτής της κρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε δουλέψει για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και στηρίζουμε και εμείς την τροπολογία Νίτρες όσον αφορά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας αυτής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλλος σκιώδης. Όχι. Κύριε Μπαλντίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Νίτες για το έργο που επετέλεσε ως εισηγητής. Νομίζω η πρόταση του είναι πλήρως αεδεκτή Και αυτό θα μας δώσει μια ευκαιρία να μην γίνει αυτό αναδρομικά και να έχει περισσότερο χρόνο η Κροατία ώστε να προσαρμοστεί όπως πρέπει σε σχέση με αυτό το νομικό πλαίσιο. Όλα αυτά βαίνουν καλώς και πολύ σωστά με καλό τρόπο παρουσιάζονται και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υποστηρίξουμε την τροπολογία αυτή στην έκθεσή του. Ευχαριστώ. Right. Μάλιστα ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, εσείς σας ευχαριστώ. Όλοι συμφωνούν λοιπόν. Πολύ καλά. Και γι' αυτό η προθεσμία θα είναι 25η Φεβρουαρίου. Αν υπάρχουν τροπολογίες. Θα τις συζητήσουμε στις 17 και στις 18 και θα περάσουμε στην περίοδο Συνόδου Απριλίου 2 προς έγκριση. Όλα τα άλλα μια και αναβλήθηκαν τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε διάφορα και μπορώ να σας υπενθυμίσω απλά και μόνο ότι έχουμε αυτή την πέμπτη μια συνεδρίαση ε, ε, από τις 9 ε, στις 10 και μισή και θα έχουμε και το θέμα της επόμενης Δευτέρας στο Στρασβούργο στην περίοδο Συνόδου και την πέμπτη επίσης έχουμε το άλλο ίμιση της ε, ψήφισης ε, ε, σε σχέση με την καταπολέμηση πλησίματος χρήματος και με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Την πέμπτη εντάξει. Meeting closed. Η συνεδρίασή μας σας ευχαριστώ.